Έκθεση της κυρίας Στάινρουκ. Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Παρακαλώ την να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καταρχάς θα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και οδησιητές για την πολύ σημαντική, καλή, εντατική συνεργασία που ε, μου προσέφεραν ευθύς εξ αρχής έχουμε νομίζω καταφέρει από κοινού μια, από μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαμορφώσουμε μια καλή και γερή έκθεση, μια βάση και θέση για τις διαπραγματεύσεις του τριμερή διάλογο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή αλλά και την Κυπριακή και Ιρλανδική Προεδρία γιατί συζητήσαμε πολλές φορές, ε, μερικές φορές να ήταν τόσο εύκολα όλα αλλά πάντως καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολύ καλές και αποδεκτές συμβαστικές λύσεις. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό έχει τρία αυτόνομα προγράμματα μεταξύ τους, καταρχάς το Progress, το, την ανάπτυξη και το συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς και για τις συνθήκες εργασίας. Το δεύτερο είναι το EURES, το δίκτυο αυτό που έχει ως καθήκον την ενημέρωση, την παροχή συμβουλών ε, και την υποστήριξη για κινητικότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και την προσφορά δυνατοτήτων ε, για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών της Ευρώπης. Το δε τρίτο πρόγραμμα, η μικροχρηματοδότηση επιτρέπει την ε, παροχή μικροπιστώσεων ε, για μικρές επιχειρήσεις, τις πιο μικρές επιχειρήσεις, για υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων ή για θέσπιση τους. Και έτσι μπορούν τώρα οι επιχειρήσεις να έχουν ε, τέτοιου τους μικροπιστώσεις. Η αρχική θέση λοιπόν ήταν τέτοια που διερωτηθήκαμε γιατί τόσο διαφορετικά προγράμματα να ενταχθούν σε ένα ε, και μοναδικό. Είχαμε πολλά ερωτηματικά σχετικά με το πόσο ταιριάζανε τα τρία αυτά προγράμματα μεταξύ τους. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν βλέπω και ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέμηση της ένδυας και άλλα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και δεν βλέπω ένα κοινό πλαίσιο για τα τρία αυτά επιμέρους προγράμματα. Δεν έβλεπα τουλάχιστον. Τώρα όμως έχουμε ένα νέο πρόγραμμα με νέο τύπο, με ένα πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, με καταπολέμηση της ένδυας, με κοινωνική ενσωμάτωση, με στόχευση στην ποιοτική απασχόληση, με ιδιαίτερους στόχους προώθησης μέσα στα επιμέρους αυτά τρία προγράμματα και με συγκεκριμένα κονδύλια. Επί παραδείγματι στο πλαίσιο του Progress έχουμε 50% των κονδυλίων ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της ένδυας και την υποστήριξη κοινωνικής ενσωμάτωσης. Για τη μελλοντική χρηματοδότηση των ε, εταιρικών σχέσεων του Eures ε, είχαμε πάλι κρίσιμες συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε για τις ε, παραμεθόρες περιοχές ιδιαίτερα να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το κοινωνικό ταμείο για του εργοδότες και του εργαζομένους, όμω εμείς αυτό θεωρήσαμε σφάλμα, γιατί θεωρήσαμε ότι θα οδηγούσε σε, σε διακινδύνευση και θα ε, προξενούσε τεράστιες δυσκολίε αυτέ οι εταιρικέ σχέσει τι διασυνοριακέ, ενώ ήδη υπάρχουν αρκετά καλά προγράμματα τα οποία κινδυνεύαν και να εξαφανιστούν ακόμη. Αυτέ οι διασυνοριακέ λοιπόν εταιρικέ σχέσει διαφυλάσσονται και εξασφαλίζονται χάρη στο πρόγραμμα Eures και η συνεργασία με, σε μερές επίπεδο με συνεννοήσεις και συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών για την προσφέτεια των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι ε, εξασφαλισμένη. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κοινό πλαίσιο με αιτήσια προγράμματα εργασίας τώρα πλέον για όλα τα υποπρογράμματα και όχι μόνο για το πρόγκρες όπως αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όταν θα ορίζει διαφορετικές, όταν θα θέλει να ορίζει διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό θα γίνεται μόνο με πρώτερη ε, διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εδώ έχουμε ένα συμβασμό που εξασφαλίζει ένα πιο σαφή ρόλο για το Κοινοβούλιο, όχι τόσο όσο θα θέλαμε εμείς, αλλά πάντως σαφή, σαφή βελτίωση. Τι δεν επιτύχαμε. Η Επιτροπή Απασχόλησης είχε ε, συνενετικά από όλε τι ομάδε προτείνει ένα τέταρτο υποπρόγραμμα να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα με πρόσθετα κονδύλια, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη σχεδίων και έργων για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαρσίω. αλλά δυστυχώ εδώ ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τίμησε τις υποσχέσεις της, ε, παρέμειναν αυτέ λόγια κενά και δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε το συντονιστό που θα θέλαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω εδώ να αντιληφθείτε ότι θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος να προσφέρουμε υποστήριξη στην απασχόληση των νέων και με τρόπο ορατό αλλά και με τρόπο αποτελεσματικό. Ε, κατά τα άλλα όμως μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τις συμβαστικές λύσεις και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορέσαμε να προχωρήσουμε αρκετό κομμάτι του δρόμου για να ε, προωθήσουμε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την συγκήτρια. Έχετε ακόμη ένα λεπτό για τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις και τώρα παρακαλώ τον Επίτροπο Άντορ να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και όλους τους κοιόδης για την επικοδομητική τους προσέγγιση προς το θέμα αυτό. Μετά από την συνεργασία των τριών οργάνων νομίζω ότι καταλήξαμε, πετύχαμε το κοινό μας στόχο. Σε περίοδο κρίσης και δημογραφικών, τεχνολογικών και κλιματολογικών αλλαγών που επηρεάζουν την αγορά εργασία και τα συστήματα κοινωνική περίθαλψη, είναι πολύ επίκαιρη αυτή η νομοθεσία. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα καινούριο εργαλείο μαζί με το Κοινωνικό Ταμείο για να μπορέσει να προωθήσει την απασχόληση την ανάπτυξη και να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το πρόγραμμα αυτό για την κοινωνική αλλαγή και την κοινο... το... καινοτομία θα, υποστηρίξει, θα στηρίξει τις προσπάθειες των που κάνουν τα κράτη-μέλη τα ίδια για να καταπολεμήσουν την ενεργεία. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετάσχουν επίσης. Σε αυτά τα πλαίσια 100 εκατομμύρια θα διατεθούν σε πειραματικά προγράμματα για την απασχόληση των νέων και την καταπολέμηση της κοινωνικού αποκλεισμού ή των προβλημάτων των πιο των ασθενέστερων ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και συνοχή στην πολιτική αυτή και κατάλληλη χρηματοδότηση στα πλαίσια της πολιτικής του 2020 καθώς και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έτσι συμπληρώνουμε τα τρία προηγούμενα προγράμματα, το ένα για την ε, απασχόληση, το άλλο το Γιούρες και τρίτον την ε, δυνατότητα μικροχρηματοδότησης. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανεργία των νέων και στην εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση της και του κοινωνικού αποκλεισμού συλλέγοντας πληροφορίες και διαδίδοντάς τες καθώς και πραγματοποιώντας διάφορες δοκιμές. Με τη συμπερίληψη του Γιούρες στο Ίζι» θα εφαρμόσουμε ειδικά προγράμματα για την προώθηση των πειραμάτων αυτών. Η κινητικότητα της εργασίας μπορεί να υποτελέσει έναν ισχυρό μηχανισμό εξισορρόπησης των προβλημάτων και των πιέσεων που αντιμετωπίζει η αγορά εργασία αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα για του νέου. Και τέλο, το εργαλείο για τη μικροχρηματοδότηση και το νέο εργαλείο για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων θα προωθήσει από το επιχειρηματικό πνεύμα και θα αποτελέσει μία βάση πειραματισμού για να δούμε τι μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μαζί με το Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το EASY θα είναι ένας ακόμη πυλώνας για την περίοδο 14 με 20 σας κατευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίτρο. Και τώρα ακούμε του εκπροσώπου των διαφορών επιτροπών με τον κύριο Λιμπεράτση πρώτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ μου δίνετε το λόγο. Είναι πολύ σημαντικά δύο θέματα για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού η διαφάνεια της χρήσης ε, και ο προορισμός των κονδυλίων. Θεωρούμε ότι καταρχάς ο ίδιος ο στόχος που είναι να δώσουμε μια νέα στην κινητικότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να μπορούν να διευκολύνονται να βρίσκουν θέσεις εργασίας, να ανταλλάζουν βέλτιστες πρακτικές και να διευκολύνεται και η κοινωνική τους ένταξη είναι οι πτυχές τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Επιπλέον, θεωρούμε ότι το να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ε, για, τον, για τα κονδύλια δεν θα είναι τόσο εύκολη. Μπορεί να έχουμε ε, λιγότερη διαφάνεια σε μικρότερα κονδύλια, αλλά ε, χρειάζονται αυτά τα χρήματα. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή μας είχαμε μόνο μία ψήφα κοτά, κάτι το οποίο καταδεικνύει την ποιότητα της εργασίας μας. Ευχαριστώ κυρία Ζούπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο παρόν πλαίσιο το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποβεί σημαντικό. Μπορεί να αποβεί σημαντικό διότι αυτό το οποίο αναζητά είναι να εδραιώσει θέσεις απασχόλησης ποιότητες ε, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τα κατάλληλα κοινωνιακά και εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχει μια καθυστέρηση αυτή τη στιγμή σε αρκετές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και ευθύνη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ελπίσουμε πραγματικά ότι θα δώσουμε μια νέα αίτηση στην ελεύθερη κυκλοφορία και δεν θα έχουμε μια υποχρεωτική μετανάστευση. Διότι κανείς δεν θέλει να χάσει τους νέους ανθρώπους ε, και το, ε, τους ανθρώπους με επαγγελματικά προσόντα τα οποία έχει εκπαιδεύσει. Μας ενδιαφέρουν επίσης οι μικροπιστώσεις και οι επενδύσεις ε, στη θετική ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι η αρχή του επιχειρηματικού πνεύματος είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, ιδίως αν ε, τελικά δεν έχουμε κατάλληλες δημόσιες επενδύσεις, όπως γίνεται με όλες αυτές τις θέσεις εργασίας που χάνονται αυτή τη στιγμή. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Κύριε piąta osoba w Europie zagrożona jest πέντε πολίτε τη Ευρώπης βρίσκεται στο κατόφλι του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι πολλοί αυτοί που ε, ε, έχουν μείνει άνεργοι. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουν οι το μέσο αυτό για τη μικροχρηματοδότηση να ξεπεράσει τα απλά λόγια και να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο χρήσιμο για τους πολίτες και να δώσει σταθερή δουλειά και απασχόληση. Χαίρομαι που αποφασίζεται να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα της πρόβλησης των νέων στην αγορά εργασίας είναι ε, η μικροχρηματοδότηση ένας πολύ σημαντικός παράγων ε, το 1 τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, θα μπορούσε να απασχολήσει ανέργους, νεαρούς ανέργους και γι' αυτό χρειάζεται αυτή η μικρό ε, χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν βέβαια και οι τοπικές ε, αρχές σε όλη αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περάμε στους μιλητές εκ μέρους των ομάδων, ο κύριος Μπουλόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Στάιμπρουκ, χάρη στην οποία μπορέσαμε να καταλήξουμε το πρώτο τέτοιο πρόγραμμα 14 με 20 που, αντιμετωπίζει διάφορε προκλήσει Η κύρια είναι να υπάρξει ένα κοινωνικό πρόγραμμα που να μπορεί να στηρίξει την αντιμετώπιση τη ανεργία και ιδιαίτερα των νέων μαζί με το συντονισμό και συνεργασία με τι χώρε μέλη. Σε αυτό το πνεύμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδυνάμωσε την ε, διάσταση της διαμεθοριακής συνεργασίας. Θέλουμε να ενισχυθεί η κινητικότητα των ζητούντων εργασία και των εργαζομένων έτσι ώστε να μπορούν μεταξύ κρατών μελών να κινηθούν για να μην φεύγουν από την Ένωση. Δεύτερη πρόκληση. Να συνενώσουμε τρία διαφορετικά προγράμματα σε ένα και μόνο χωρίς να χαθούν οι στόχοι τους. Το Κοινοβούλιο πέτυχε πρώτον η διαχείριση αυτών των προγραμμάτων να απλοποιηθεί και να υπάρξει σωστός συντονισμό και με κατάλληλο προπολογισμό. έτσι ώστε να ενισχυθούν και από τα τρία προγράμματα εκείνα που ενισχύουν την νεολαία. Τελευταία πρόκληση να επιτραπεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέχρι ενός καινούργιου συστήματος μικροχρηματοδότησης. Προσωπικά θα ήθελα να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέμα των επιχειρήσεων που θεωρούνται κοινωνικά ενάρετες. Έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί και ο κοινωνικός πειραματισμός, η καινοτομία για να έχουν έτσι τα κράτη όλα τα εργαλεία που χρειάζονται στα χέρια τους για να αντιμετωπίσουν αυτά τα τεράστια προβλήματα της ανάπτυξης και της ανεργίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέρντιν. Εδώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Η κοινωνική χρηματοδότηση της Ένωσης είναι θέμα που το συζητήσαμε πολλές φορές αυτή την εβδομάδα. Το νέο αυτό πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία θα χαράξει νέους δρόμους καινοτόμους. Πράγμα στο οποίο οφείλουμε στις προσπάθειες της ομάδας του Κοινοβουλίου και της Γιούτα Στάνιμπροκ ιδιαίτερα που θέλησε να συνενώσει τρία υπάρχοντα προγράμματα σε ένα ενιαίο με καθαρή και διαφανή χρηματοδότηση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της αύξησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού διευκολύνοντας τη μικροχρηματοδότηση, την επαγγελματική κινητικότητα όπου η Ευρώπη μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα. λόγω της τεχνογνωσίας της ή των χρημάτων που θα θελήσει να διαθέσει. Αυτά είναι και οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώς. κυρία Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που πίστεψε τόσο πολύ σε αυτό το πρόγραμμα για να γίνει ρεαλιστικό. Με απογοητεύει βέβαια το γεγονός ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν εξίσου και τα τρία προϋπάρχοντα προγράμματα. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της μικροχρηματοδότησης, το ύψος 25.000 ευρώ για όσους κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους ή για όσους έχουν δυσκολία στη δανειοληψία. Αυτά τα νέα δάνεια θα βοηθήσουν και τους ε, νέους που θέλουν να δημιουργήσουν επιχείρηση. Από το 10 και μετά πάνω από 6.000 τέτοιοι νέοι επιχειρηματίες έχουν ήδη αποφεληθεί με το, από το πρόγραμμα Microfinance. Μάλιστα από τότε είχα πάρει και εγώ μέλος στους τριμερείς διαλόγους και χαίρομαι ιδιαίτερα που το πράττω και σήμερα. Η Ιρλανδία, η χώρα μου δηλαδή, έχει πρόσβαση σε, αυτό το εργαλείο γιατί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι τεράστιο πρόβλημα για τους νέους ιδιαίτερα όταν έχουν κοινωνικά προβλήματα για τη δημιουργία των επιχειρήσεών των το ταμείο αυτό δεν θα τα λύσει βέβαια όλα, αλλά παρόλα αυτά θα βοηθήσει στην αυτοαπασχόληση και στην δημιουργία επιχειρηματικού πνεύματος. Ξέρω ότι είμαι βέβαιο ότι οι Ιρλανδοί επιχειρηματίες θα το δεχτούν με χαρά. Επίσης χαίρομαι διότι βλέπω ότι το Γιούρες είναι στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας και ότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα one-stop shop έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να παρακολουθούν πιο εύκολα τις ε, ροές της κινητικότητας και να αντιμετωπίζουν τα πιθανά προβλήματα. Ευχαριστούμε κυρία Σρότερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Κοινοβούλιο μέσα σε αντίξωε συνθήκε. κατάφερε να διαπραγματευτεί μια καλή συμβαστική λύση που θα την υποστηρίξουμε. Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για τη ε, διατήρηση της υποστήριξης για τις περιοχές Γιούρες. Ε, μπόρεσε το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ένα 18% από τα 920 συνολικά εκατομμύρια ευρώ για τις ε, παραμεθόριες περιοχές, για τις διασυνοριακές ε, ε, συνεργασίες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διατηρούνται αυτές οι δυνατότητες για τα επόμενα 7 χρόνια και δίνεται να αναπτυχθούν και νέες εταιρικέ σχέσεις πέραν των συνόρων. Αυτό αποτελεί μια καλή είδηση πιστεύω και για τις εταιρικέ σχέσεις γιούρες και για όσους μένουν κοντά στα σύνορα για ταξιδεύουν από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο των Διασυνοριακών Εταιρικών Σχέσεων απερίφθησαν από, την, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα οδηγούσαν σε απόλυτη απαξίωση τους και αποτυχία τους. Θα έπεφταν δηλαδή σε εθνικές, στην εθνική αρμοδιότητα και δεν θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθούν προγράμματα για διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. Οι παραμεθόριες περιοχές ωστόσο ε, γνωρίζουν πάρα πολλούς υπερμεθοριακούς εργαζομένους, μένουν στο ένα κράτος, εργάζονται στο άλλο και πρέπει και να ενημερώνονται ε, για τα δικαιώματά τους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το κοινωνικό ε, σύστημα, της κοινωνική, την κοινωνική νομοθεσία όπως ισχύει και αυτό μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να εξασφαλιστεί. Επιτρέψτε μου να κάνω μια ακόμη παρατήρηση πολύ σημαντική για το μέσο για την μικροχρηματοδότηση και εδώ έχει επιτύχει ένα μεγάλο, μια μεγάλη νίκη το Κοινοβούλιο με τους αγώνες του διότι εξασφαλίζει την χορήγηση αυτών των μικροεπιχορηγήσεων ε, και σε ιδιώτες αλλά και σε μικρές επιχειρήσεις που δεν είχαν καμιά άλλη δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά σε πολύ μικρές, ε, για πολύ μικρά ποσά, πραγματικά πολύ μικρά ποσά, αυτές οι μικροπιστώσεις μπορούν να χορηγούνται σε προγράμματα μόνο πιλωτικά και γι' αυτό θα θέλω να απευθύνω έκκληση προς όλα τα κράτη-μέλη από τη θέση αυτή να κοιτάξουν και από πλευρά του πρόγραμμα, στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να αναπτύξουν και άλλες μικροπιστώσεις για να συμπληρώσουν αυτό το μέσο. Γιατί μόνο έτσι θα είναι δυνατόν να... οι ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά, σε πιστώσεις δηλαδή από την ελεύθερη αγορά, να εξασφαλίσουν ε, τη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις τους, για την ίδρυση της νέας επιχειρήσης ή για την διέξοδο από την ανεργία. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα καλό, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να στεφθεί με επιτυχία και πιστεύω ότι στην απόφαση του Κοινοβουλίου έπαιξε εδώ πολύ πολύ σημαντικό ρόλο και έδωσε μια νέα σημαντική ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ευχαριστώ πολύ. Φάνταν Κάμεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πολίτες καθημερινά διαπιστώνουν τις συνέπειες των ε, εσφαλμένων, ε, των ε, κοντόφθαλμων ευρωπαϊκών πολιτικών και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές κατά την άποψή τους υποβάλλει παρανοϊκές προτάσεις, ε, οι οποίες έχουν προκύψει από θεωρητικά εγχειρίδια. Νομίζω ότι πρέπει οι πολίτες να προσεγγίσουν την ε, ε, πολιτική και να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο και να μπορούν να διαμορφώσουν οι την πολιτική τους και θεωρούν ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να καθορίζουν αυτές τις προτεραιότητες και όχι να αφήνουμε το ελεύθερο σε δογματικές ε, αποφάσεις των Ευρωπαίων ε, γραφειοκρατών. Τα πειράματα αυτής της μορφής θα έπρεπε να σταματήσουν και θα πρέπει να αλλάξουμε σελίδα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, να τα στείλουμε πλέον στις χώρες μέλη και να μην σπαταλούμε χρήματα για αυτούς τους ανόητους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι κάνουν. Ευχαριστώ η κυρία Ρεγκίνα Μπάστος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Άντορ για την παρέμβασή του. Η κρίση την οποία βιώνουμε ε, δημιούργησε κοινωνικά προβλήματα και για την απασχόληση και διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των ε, πιο σημαντικών κρατών είμαστε ένα σύνολο, αλλά τα προβλήματα σε μία χώρα μέλους μπορεί να δημιουργήσουν συνέπειες και σε άλλη χώρα μέλος και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει και ο κατάλληλος συντονισμός και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όσον αφορά την εργασία και όσον αφορά την καταπολέμηση της άνδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για τη μάχη που δίνονται για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε τους κοινωνικούς στόχους που περιλαμβάνονται στη στρατηγική 2020. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα προγράμματα όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και επίσης ε, ε, μέσω αυτό να έχουμε σημαντικά προγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και να τα στα προβλήματα. Το Progress, το EORES και το πρόγραμμα της μικροχρηματοδότησης ε, για θέματα απασχόλησης δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η κατάσταση για τις χώρες που έχουν πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας και κυρίως ανεργίας για τους νέους είναι πολύ σοβαρή. Και θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό, διότι θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της λύσης και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα ε, δίνουν κίνητρο για την ε, πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία και θα βοηθήσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες. Ευχαριστώ κυρία Στρέλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια, την κυρία Στάινμπουργκ, για την εξαιρετική της έκθεση. Να ευχαριστήσω επίσης διότι υποστήριξε τις προτάσεις της Επιτροπής Γυναικών. Η διάσταση του φύλου είναι μία από τις ε, αναπόσπαστες πτυχές των εργασιακών πολιτικών και των ε, θεμάτων απασχόλησης. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα νέα μοντέλα εργασίας και τους κινδύνους που υπάρχουν για την υγεία και την ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να μπορέσουμε να συμφιλειώσουμε την οικογενειακή και την εργασιακή ζωή και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας ε, ε, θα πρέπει να διέπονται και από τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την βοήθεια στην οικογενειακή ζωή, να υπάρχουν άδειε, για παράδειγμα ναι, και ναι, ναι. Ε, γονικές και για άνδρες και για γυναίκες και θα πρέπει ε, να τονίσουμε το θηλυκό στοιχείο στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση για να επιτύχουμε αυτό το στόχο του 75% απασχόλησης των γυναικών όπως προβλέπει η Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ η κυρία Σάγια. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Στην Επιτροπή κάναμε πολύ καλή δουλειά υπό την καθοδήγηση της εισηγητρίας. Οι, δου... οι θέσεις εργασίας του τους χρειάζονται και νέες αρμοδιότητες και για την απόφαση να ε, μετακινηθούμε για να βρούμε μια θέση εργασίας. Λίγοι είναι αυτή τη στιγμή ακόμη οι Ευρωπαίοι που εργάζονται ε, και κατοικούν σε διαφορετική χώρα. Υπάρχουν προβλήματα τεχνικά οι μεγαλύτερα πραγματολογικά στοιχεία όπως η παγκοσμιοποίηση, η γέννηση του πληθυσμού, τα ζητήματα της ενέργειας, τα οποία διευκολύνουν όμως τώρα τις ε, ταχείες μεταλλαγές σε διαφορούς τομείς. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, ε, το πρόβλημα είναι αυτό της ανεργίας ενώ θα μπορούσε να προσφέρει θέση απασχόληση για τους πάντες η Ευρωπαϊκή Ένωση και αηφορία βιωσιμότητας της εργασίας, αλλά αυτό χωρίς βεβαίως να ε, χωρίς τα προγράμματα αυτά δεν θα μπορούσε να το προωθήσει. Θέλουμε προγράμματα λοιπόν τα οποία θα λειτουργήσουν και θα ενισχύσουν τις εργασίες. Ιδιαίτερα το, το, το δίκτυο Eures πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο χάρη στα πιλωτικά προγράμματα το Γιούρες Απασχόληση όπως ονομαζόταν στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν μια διάσταση πολύ σημαντική που ενεθάρρυνε τους νέους να αναζητήσουν τα εργασία στο εξωτερικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ε, δυνατότητες τώρα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου προς τον εισηγητή. Εδώ στηριζόμαστε σε τρία εφιστάμενα προγράμματα για ένα νέο πρόγραμμα. Προγράμματα τα οποία ενισχύουν τι ε, τις, ευκαιρίες, τις ευκαιρίες στην κοινωνική ενσωμάτωση, την καταπολέμηση ανεργίας μέχρι 25.000 ευρώ δάνειοδότηση για μικρές επιχειρήσεις, μικροχρηματοδότηση δηλαδή όπως είχαμε και στην Ισλανδία τελευταία χρόνια. Χάρη στο Eures θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε καλύτερα τις ανάγκες των εργαζομένων με, τους, ε, με των εργοδοτών. Έχουμε ε, πολύ σημαντικά ποσοστά ανεργία στη χώρα μου, την Ιρλανδία, που με ανησυχούν πρέπει να πω, όλα από τα άλλη θεωρώ ότι όποιο νέο θέλει να ταξιδέψει για να αναζητήσει ναι. εμπειρίε σε μια άλλη χώρα θα πρέπει να έχει καλή ενημέρωση και ευκαιρίε για απασχόληση. Σε αυτό συμβάλλει το Eures. θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για τα όσα επέτυχε. Το 20% των 500 εκατομμυρίων που είχαν προβλεφθεί για τη διάσταση Progress. Ιδιαίτερα θα πρέπει να πάνε στην απασχόληση των νέων και τη δυνατότητα για την μικροχρηματοδότηση που θα προσφερθεί στις μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα η υποστήριξη θέσης εργασίας και κοινωνικές πολιτικές οι οποίες δεν θα αποκλείουν κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο... Δεν βλέπω να στείλει κανείς λόγο τώρα. Παρακαλώ εσείς. Ο κύριος πάρει ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κοινωνική οικονομία συνεχίζει να αυξάνεται ακόμη και μέσα στην κρίση. Στη χώρα μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες καινούργιες μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις στο ΣΥΡ ας πούμε που προσφέρουν υπηρεσίες στους πιο αδύναμους. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού πρέπει νομίζω να προσεχθεί από την Κομισιόν να γνωρίζει καλά τι σημαίνει κοινωνική επιχείρηση και η χρηματοδότηση, η μικροχρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Βρετανία λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Μέσω οργανώσεων που θα τις ελέγχουν οι ίδιοι ή μη προνομιούχοι. Ξέρουμε ότι τα αρχικά του προγράμματος αυτού λέγονται easy, αλλά ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η επιτυχής εφαρμογή του. Ευχαριστούμε ο Επίτροπος Άντορ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την υποστήριξή σας στο νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο και ιδιαίτερα την κυρία Στάινμπρουκ που έκανε τέτοια προσπάθεια για την σωστότερη εφαρμογή του προγράμματος αυτού και πρόσεξε όλες τις λεπτομέρειες πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί παρά τις μικρές περικοπές που ε, συνέβησαν αυξήθηκε η ποιότητα του προγράμματος και νομίζω ότι με αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε επιπτώσεις θετικές να αποτελέσει δηλαδή ένα πραγματικό εργαλείο για την πραγματοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020 μόνο όμως εάν πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της κοινωνικής καινοτομίας την ε, αντιμετώπιση του προβλήματος των, μεταναστε, των μεταναστών που θα μπορούσε να παίξει, όπως έχει ήδη παίξει, πολύ θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά πολέμηση της ανέχειας και της ανεργίας. Η γενετικότητα επίσης είναι πολύ σημαντική για την ε, αγορά εργασίας της Ευρώπης και σε 5-10 χρόνια θα γίνει ακόμα πιο σημαντική. Το Γιούρες πρέπει να ενισχυθεί και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ζητήσαμε και εμείς την ενδυνάμωσή του και βλέπω με ικανοποίηση ότι και εσείς το δέχεστε. Χαίρομαι επίσης που υποστηρίχθηκε τόσο πολύ η μικροχρηματοδότηση ιδιαίτερα από την πλευρά της Ιρλανδίας από την κυρία Χάρκιν, την κυρία Κοστέλο γιατί είναι πολύ σημαντικό και για εκείνη και για το Ηνωμένο Βασίλειο η δυνάμωση αυτή της κοινωνικής οικονομίας. Αυτά βέβαια πρέπει να συνεχίσουν και στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Όλες οι χώρες μέλη έχουν υποφεληθεί από το εργαλείο της μικροχρηματοδότησης και θα ήθελα οι χώρες που δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη να το ξανασκεφτούν, να θελήσουν να συμμετάσχουν και εκείνες. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα επιτυχιών του προγράμματος αυτού που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν ως πρότυπο και έμπνευση. Τώρα, η εφαρμογή του EASY θα είναι βέβαια ευθύνη της Κομισιόν και ελπίζω ότι κατά την εφαρμογή του θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση με την εισηγητρία, την κυρία Στάινρουκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Θα ήθελα για όσους εξέφρασαν ε, επικρίσεις να είχαν συνεργαστεί στα προγράμματα αυτά για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών στις χώρες τους για να έχουμε καλές θέσεις εργασίας, για να βοηθήσουμε αυτούς που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση, για να στηρίξουμε τους νέους στην αναζήτηση μιας θέσης εργασίας. Και είχε δίκιο κύριε Επίτροπε, επιτύχαμε το στόχο μας όσο και αν ήθελα περισσότερα κονδύλια, που όμως δεν ήταν στο χέρι μου. Νομίζω ότι μπορεί, μπορούμε έτσι να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο την κοινωνική Ευρώπη και ευχαριστώ όλους όσους με υποστήριξαν. Και εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Η ψηφοφορία αύριο στο 12 το μεσημέρι. Και τώρα το τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης. Η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Την ερώτηση